Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier. Cari colleghi, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα μου επιτρέψετε να καλωσορίζω στην σημερινή μας Ολομέλεια τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας εδώ είναι μεγάλη τιμή για μας το ότι επιλέξατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δεύτερη έξοδό σας από την Γερμανία στα πλαίσια του νέου σας ρόλου μετά από αυτήν στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα και μόνο ούτε τρεις εβδομάδες από την ημέρα που αναλάβατε τη νέα σας θέση. Η παρουσία σας εδώ λοιπόν δείχνει την αφοσίωσή σας στην Ευρώπη την ισχυρή αποφύωση. Σας ζητήσατε περισσότερο θάρρος για την Ευρώπη, για μια καλύτερη Ευρώπη, ελεύθερη Ευρώπη, Ευρώπη εργασίας, ευημερίας και δικαιοσύνης. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι το θάρρος το οποίο αναζητείτε μπορείτε να το βρείτε ανάμεσα στα μέλη αυτού εδώ του Κοινοβουλίου. Με την παρουσία σας λοιπόν κύριε Πρόεδρε υπενθυμίζετε και την αφοσίωση της χώρας σας για την Ευρώπη, μια πολύ σημαντική προσπάθεια, ιδιαίτερα μετά από την απόφαση ενός κράτους μέλους να εξέλθει της Ενώσεως. Βιώνουμε δύσκολες στιγμές, έχουμε ζήσει αντίστοιχες στιγμές και στο παρελθόν και πάντα η πολιτική μας ένωση βρήκε την κατάλληλη λύση με τα κατάλληλα μέτρα Αγαπητέ Πρόεδρε, δεν θα σας ζητήσω να δώσετε λεπτομερείς απαντήσεις σήμερα, αλλά θα σας ζητήσω να εργαστείτε μαζί μας για το κοινό μας μέλλον. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την παρουσία σας κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Αντώνιο, αγαπητοί βουλευτές, ε, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητέ Ζαν Κλοντ, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά χαρά και τι